Good Κυρίες και κύριοι, αγαπητές συνάδελφοι, την προσοχή σας παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 27 της ημερησίας διάταξης σχετικά με τις ε, συνθήκες εργασίας και πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία των Παγκλαντές στα πλαίσια των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, κάποια ατυχή γεγονότα στην ε, βιομηχανία μετισμού στον Μπαγκλαντές έχουν ευστήσει την προσοχή μας στις συνθήκες εργασίας στον Μπαγκλαντές πυρκαγιές ε, σε εργοστάσια και κατάρρευση κτηρίων ε, αρκετών εκτερίων, Να σας υπενθυμίσω ότι το Μπαγκλαντές επωφελείται από μεταχείριση μηδενικών δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το καθεστώς Everything But Arms, οτιδήποτε πλην όπλων. Αλλά το Μπαγκλαντές είναι ένα σημαντικός Τέλος, το 90% των εξαγών των Παγκλαντές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμα ενδύματα, ενώ το 60% των εξαγών των έτοιμων ενδυμάτων από τον στέλνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τεράστια ευθύνη για να παρακολουθεί τα γεγονότα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασία των Μπαγκλατέ. Γι' αυτό με μεγάλη ικανοποίηση θα καλωσορίσω στη συνεδρίαση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κυρία Ισμάτ Γιαχάν, η οποία είναι πρεσβευτή ε, του Μπαγκλατέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια ανταλλαγή απόψεων για τις συνθήκες εργασίας στη χώρα της στα πλαίσια των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Παγκλαντές, καθώς και τον κύριο Χουάνμπονγκ, ο οποίος είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Και θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Φραντσέσκο Μάρκη, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής του Ρετσέξ, και τον κύριο Λόρεντς Μπερτσάλ, ο οποίος είναι διευθυντής της Fair Trade Association. Νομίζω ότι θα έχουμε μία καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα ξεκινήσω. δίνοντας το λόγο στην αξιότιμη πρεσβευτή του Μπαγκλαντές. Και πάλι καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Μορέιρα, αξιότιμοι βουλευτές, κύριε Αναπληρωτή Διευθυντή της ILO, της Γενικής Διεύθυνσης ε, Eurotex και κυρίες και κύριοι. Η παρουσία μας σήμερα δείχνει την ε, ε, συλλογική μας δέσμευση να αυξήσουμε τα πρότυπα ασφαλείας στις, στους χώρους εργασίας στον Παγκλατές. Πρόσφατα, μετά την κατάρρευση εργοστασίου τον Απρίλιο και μετά από την πυρκαγιά στο Ταζρίν. Έχει επικεντρωθεί η προσοχή του κόσμου στην ε, βιομηχανία ρούχων του Μπαγκλατές ε, και πιο συγκεκριμένα έχει ε, επικεντρωθεί η εξέταση του κόσμου στο θέμα αυτό και αυτό το επικροτούμε. Μπορεί να ακούγεται κοινικό κάπως, αλλά από αυτές τις τραγωδίες είδαμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Ε, την ε, συνειδητοποίηση ότι πρέπει να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση. Μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα, οι φίλοι και εταίροι μας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένοι τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, που είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος και άλλοι μας έχουν θυμίσει ότι πολλά απομένουν να γίνουν όσον αφορά τα πρότυπα ασφαλεία και τις εργασιακές συνθήκες. Και είναι επίγον ε, να ε, δούμε αποτελέσματα. Δύο ψηφίσματα υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 ε, Ιανουαρίου και 23 Μαΐου αντίστοιχα του 2013 που τονίζουν ακριβώς τα ζητήματα αυτά. Οι ευρωβουλευτές καλούν τις πολυεθνικές ε, μάρκες ε, να ε, ακολουθήσουν τις πρακτικές εταιρική ευθύνη και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιριών ε, που λειτουργούν στο εξωτερικό. Ε, κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζουμε ότι η ραγδαία ανάπτυξη του, της βιομηχανίας ε, ρουχισμού και η πρακτική υπεργολαβία, της υπεργολαβίας έχει οδηγήσει στην ύπαρξη εργοστασίων τα οποία δεν συμμορφώνονται πάντα με τα πρότυπα ασφαλείας. Και εδώ συμμεριζόμαστε την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει να ληφθούν επίγοντα διορθωτικά μέτρα. Να σας θυμίσουμε ότι ε, λίγες εβδομάδες μετά την ε, κατάρρευση του Ράνα Πλάζα, ε, ο Υπουργός Εξωτερικών του Μπαγκλαντές ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για να ενισχύσει τη δέσμευση του Μπαγκλαντές και να έχει συναντήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι και έχουμε συνεχίσει τη στενή μας συνεργασία ε, με τους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καθώς ε, και με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Πιστεύω ότι βασικό επίκεντρο σήμερα είναι να δούμε πώς, τι αποτελέσματα έχουν επιφέρει οι κοινέ μας προσπάθειες και επικροτώ την προσπάθεια αυτή να μοιραστώ μαζί σας κάποιες δράσεις που ήδη έχουμε αναλάβει και να δούμε πού βρισκόμαστε και πού μπορούμε να πάμε. Καταρχάς, να είμαι σαφής ότι η κυβέρνηση του Παγκλατές είναι απόλυτα δεσμευμένη ε, ε, να επιφέρει ε, σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τα πρότυπα ασφαλείας και τα εργασιακά δικαιώματα στην χώρα. Η Ένωση Βιομηχανιών επίσης έχει αναλάβει δράση αμέσως μετά το ε, περιστατικό του Σαβάρ ε, ε, έχουμε αναλάβει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες μεταξύ άλλων την σύλληψη των ιδιοκτητών του κτηρίου και την δίωξή τους για να συμπληρώσουμε κάποια κενά που υπάρχουν. Ε, υιοθετήθηκε μία τριμερή κοινή διακήρυξη στις 4 Μαΐου σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο εργασία στην ΤΑΚΑ και ακολουθήθηκε αυτό από ένα τριμερέ εθνικό σχέδιο δράση. Ε, επίσης, ένα σύμφωνο βιωσιμότητα υιοθετήθηκε στην Γενέβη στις 8 Ιουλίου. Με την ε, συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών του Μπαγκλατές, τον ε, Επίτροπο Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τον Γενικό ε, Διευθυντή του ILO. Και τα βασικά στοιχεία αυτού του συμφώνου είναι τα εξής. Τροποποίηση του εργασιακού νόμου του 2006. Δεύτερον, πρόσληψη 200 επιπλέον επιθεωρητών εργοστασίων μέχρι το τέλος του 2013. Τρίτον, εξέταση όλων των ε, κτηρίων των εργοστασίων μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Σύντομα να αναφερθώ στις ε, δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει μέχρι στιγμής. Ε, ο εργασιακός νόμος του 2006 τροποποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου και έχουμε συμπεριλάβει τώρα κάποια τμήματα που επιτρέπουν μεταξύ άλλων στους εργάτες διαβριμένα δικαιώματα ε, συλλογικής δράσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και μέχρι το τέλος ε, του 2013 καταβάλουμε προσπάθειες ώστε οι τροπολογίες αυτές ε, να εφαρμοστούν στην πράξη. Στο νέο νόμο Ε, προβλέπεται να ε, ε, υποχρεωτικά ένα κέντρο υγείας στα εργοστάσια με πάνω από 5.000 εργαζομένους και επίσης Υπουργική Επιτροπή Εργασίας έχει δημιουργηθεί με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες των εργαζομένων στις ζώνες μεταποίησης. Επίσης, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την ε, εκπαίδευση, πρόσληψη ε, και τοποθέτηση επιθεωρητών ε, και το Υπουργείο Εργασίας ήδη έχει, έχει διορίσει επιθεωρητές και άλλοι 200 θα προσληφθούν σύντομα. Επίσης, τελικά, η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να έχει 800 επιθεωρητές. Επιπλέον, Υπάρχουν άλλες ε, κυβερνητικές αρχές που ασχολούνται με θέματα ε, ασφαλείας, όπως είναι η πυροσβεστική, η αρχή ανάπτυξης ε, κεφαλαίου, της καθώ καθώς και της περιοχής Ψητακών. Και στόχος είναι να ενισχυθούν η υποδομή και η οργάνωση. Με τον νέο εργασιακό νόμο, οι ιδιοκτήτες εργοστασίων θα πρέπει να ε, παρέχουν ε, εξοπλισμό ασφαλείας ε, και σωστή εκπαίδευση. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και των πολυεθνικών εταιριών και λιανοπολιτών που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν τις αιτίες των καταστροφών που είδαμε στο πλαίσιο του Εθνικού Τριμερούς Σχεδίου που περιλαμβάνει αξιολόγηση 3.500 εργοστασίων ε, ρούχων ε, στην χώρα. 30 ομάδες ε, με επικεφαλής το, πανεπιστήμιο, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μπαγκλαντές και εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα ξεκινήσουν την επιθεώρηση των εργοστασίων ρουχισμού αυτών τον μήνα. θα ε, εξετάζουν ε, αν υπάρχουν δομικά προβλήματα και θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων. 2.000 τέτοια εργοστάσια θα επιθεωρηθούν μέσα σε τρει μήνες. Επιπλέον, η Συμφωνία για ε, τη, ε, την ασφάλεια κτηρίων ε, κάποιων ευρωπαϊκών και, και αμερικανικών εταιριών θα επιθεωρήσει ανεξάρτητα περίπου 750 με 1000 εργοστάσια, καθότι οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν από τρεις ε, διαφορετικούς φορείς, ε, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ε, συντονιστούν οι διάφορες πρωτοβουλίες και να υπάρξουν κοινά πρότυπα. Το Υπουργείο Εργασία συνεργάζεται με του φορεί αυτού για να συντονίσει τι προσπάθειε ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη εργασιών και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοβουλειών. Για να υπάρξει επιτυχημένο συντονισμό ε, σημαντικό είναι να συμμετέχουν και εθνικοί φορείς ε, στην διευθύνουσα ομάδα ε, της του Συμφώνου για την Ασφάλεια των Κτηρίων των Ευρωπαϊκών Εταιριών. Πιστεύω ότι αν συνεργαστούν στενά όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κτηρίων με αποτελεσματικό τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, να σας θυμίσω ότι το Consortium για τα Δικαιώματα των Εργατών, ε, που είναι ε, ανεξάρτητος ε, φορέας παρακολούθησης, έχει υπολογίσει ότι χρειάζονται περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια ώστε να συμμορφωθούν όλα τα εργοστάσια με τις απαιτήσει. Μπορεί αυτό το ποσό να φαίνεται τρομακτικά υψηλό, εάν όμως το μοιράσουμε σε 5 χρόνια, μόνο 10 cents παραπάνω θα χρειαστούν για καθένα από τα 7 δισεκατομμύρια ε, ε, τεμάχια ρουχισμού που θα ε, εξαχθούν. Πιστεύω ότι οι καταναλωτές στη Δύση είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ε, μία ε, μικρή αύξηση ε, για τα εκατομμύρια γυναικών που ράβουν τα ρούχα τους σε μακρινές χώρες. Θα καλωσορίσουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διασφαλιστεί η δίκαιη τιμολόγηση. Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια επιτροπή για να επανεξετάσει το, τους ελάχιστους μισθούς για ε, τους εργαζομένους στον τομέα του ρουχισμού, αλλά και υπάρχουν προτάσεις ε, και από τους εργοδότες και από τους εργαζομένους ε, και ελπίζουμε να υπάρξει συνένεση τελικά. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να πω ότι εάν Εκτός ε, εάν ε, πετύχουμε δίκαιη τιμολόγηση, οποιαδήποτε ε, αύξηση στην αμοιβή των εργαζομένων δεν θα έχει νόημα στο ανταγωνιστικό, δεν θα είναι δυνατή στο, στο ανταγωνιστικό διεθνές εμπόριο. Ζητάμε από τους βιομηχάνους ε, να ε, κάνουν αυτό που πρέπει. Σημαντικό όμως είναι και οι εισαγωγείς και οι αγοραστές να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Ένα ε, κοινωνικό πλαίσιο θα πρέπει να αναπτυχθεί όπου και οι λιανοπολιτές να συμμετέχουν. Και για να πούμε και κάτι θετικό, μας έχει ενθαρρύνει η διάθεση κάποιων σημαντικών ε, εταιριών στον τομέα αυτών. Ελπίζουμε ότι και οι άλλες ε, πολυεθνικές εταιρείες θα ακολουθήσουν τις προσπάθειες αυτές στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ήδη αναφέρθηκα στην αποζημίωση που ε, δόθηκε μετά από τα τραγικά περιστατικά που ανέφερα έχει δοθεί αποζημίωση από το Κυβερνητικό Ταμείο ε, στις ε, οικογένειες ε, των θυμάτων. Μπορεί να μην ανέρχεται στο ύψος που θα θέλαμε όλοι, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι από πλευράς της κυβέρνησης καταβάλλονται ακόμα προσπάθειες. Να σας θυμίσουμε επίσης ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Γενέβη ε, είχε οργανώσει μια διάσκεψη η Industrial Global Union όπου συμμετείχαν 9 από 29 ευρωπαϊκές μάρκες για να συζητήσουν ε, τις ε, μακροπρόθεσμες, έναν μακροπρόθεσμο μηχανισμό αποζημίωσης για τα θύματα της Εράνα Πλάζα και του Ταζρίν. Είδαμε ότι υπήρχε επιφύλαξη αρκετών εταιριών να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο μηχανισμό αλλά η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα ε, έτοιμου ρουχισμού ε, απαιτεί ε, την δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών, την μεταφορά των ιδιαίτερα ευάλωτων εργοστασίων. Το πρώτο τέτοιο χωριό έτοιμου ρουχισμού δημιουργείται και δημιουργούνται και ε, χώροι για να διαμένουν ε, οι γυναίκες ε, που εργάζονται εκεί. Κύριε Πρόεδρε, ο τομέας έτοιμου ρουχισμού αποτελεί το βασικό μέρος των εξαγωγών μας προς την Ευρώπη, όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας απασχολεί 4 εκατομμύρια ανθρώπων, κυρίως γυναίκες, σε πάνω από 5.000 εργοστάσια. 20 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από την βιομηχανία αυτή. Υπάρχουν ε, σχετικές ε, βιομηχανίες όπως είναι η συσκευασία, η βαφή των ρούχων κλπ. Ε, και έτσι ο αντίκτυπος του τομέα αυτού είναι ακόμα μεγαλύτερος τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες ο βιομηχανικός αυτός τομέας έχει συμβάλει στην πολύ σημαντική ε, κοινωνική αλλαγή στην χώρα μας. Ε, έχει στηρίξει ιδιαίτερα τις γυναίκες από τα πολύ φτωχά νοικοκυριά. Ε, και ο γενικός αντίκτυπος δεν μπορεί καν να μετρηθεί. Εάν θέλουμε να έχουμε έναν βιώσιμο τομέα έτοιμου ρουχισμού στον Μπαγκλατές που να ε, ε, στηρίζει τη ζωή 4 εκατομμυρίων γυναικών ε, και των εξαρτώμενων οικογενειακών μελών τους, θα πρέπει να διασφαλίσουμε βιώσιμη πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ενισχύσει και την σχέση ανάμεσα στο εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη. Η διευκόλυνση του EPA προς τον Μπαγκλαντές ε, είχε ε, σημαντικό αντίκτυπο στον κοινωνικο τομέα της χώρας, ε, στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας και αυτό αναφέρεται συχνά ως επιτυχία του EPA σε μια από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες το 20% του ε, πληθυσμού του Μπαγκλαντές ε, θεωρείται ε, ότι είναι πληθυσμός μιας από τις ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες. Ωστόσο, το Μπαγκλαντές δεν θεωρεί δεδομένη την βοήθεια αυτή που του δίνεται. Θυμίζω την δήλωση του Επιτρόπου Καρέλ Δεκούχτ ότι ξεκινάμε ένα ταξίδι μαζί, το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Σημείωσε ότι θα είναι σημαντική πρόκληση για τον Παγκλατές και ε, ότι γνωρίζει την ανάγκη του Παγκλατές να λάβει ε, ενίσχυση και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να βοηθήσει. Ε, αυτό μας παρηγορεί. Πιστεύουμε ότι αυτό το ταξίδι είναι συλλογικό. Είμαστε αποφασισμένοι να οικοδομήσουμε εταιρική σχέση και να ε, τις αναπτύξουμε περαιτέρω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, μας έχει δώσει την υποστήριξή του και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, συνεχίσει τις προσπάθειες, μας, τις προσπάθειες μαζί μας σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Το Μπαγκλαντές, όπως και οποιαδήποτε άλλη τουρκική δημοκρατία, ε, θα πρέπει να εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις ε, για να υπάρξει ευρεία συνένεση, κάτι που κατά καιρού μπορεί να φαίνεται ιδιαίτερα δαπανηρό από πλευράς χρόνου. Αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως χαλάρωση καθυστέρηση από πλευράς της κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, να ε, διαβεβαιώσω και εσάς και όσους ενδιαφέρονται ε, για την κατάσταση των εργοστασίων στον Παγκλατές ε, ότι το Παγκλατές συνεχίζει ειλικρινά να καταβάλει προσπάθειες και είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τις προσπάθειες μαζί με όλους τους ενδιαφορομένους ώστε να αντιμετωπιστεί το δύσκολο θέμα των προτύπων ε, ασφαλείας και εργασίας στον τομέα ρουχισμού της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρέσβη. Ήρθε η ώρα τώρα να ακούσουμε την άποψη των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκινώντα από την εισηγήτρια για την Νοτιοανατολική Ασία, ε, τον εισηγητή για την Νοτιοανατολική Ασία, τον κύριο Μέρφυ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρέσβη. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκάθαρα διατυπώσει τη θέση του σε σχέση με την τραγωδία, την πυρκαγιά στο ε, εργοστάσιο και την κατάρρευση του εργοστασίου στην ε, Πλάζα. Εκφράσαμε την λύπη μας ε, τον, για τις ανθρώπινες απώλειες, καθώς επίσης και την ανάγκη να αλλάξουν τα πράγματα. Και πράγματι έχουν, έχουμε δει κάποια σημάδια ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί η άσκηση πίεσης από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά επίσης και από την κοινωνία των πολιτών στο Μπαγκλαντές. Έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η αλλαγή θα είναι πραγματική, θα επέλθει στην πραγματικότητα και θα διαρκέσει. Έχω ε, ερωτήσεις. Ένα από τα ζητήματα που με εξέπληξε είναι αυτό το συνολικό κόστος που αναφέρατε, ε, που θα είχε ε, προκειμένου που θα, θα έπρεπε να αναλυθεί και προκειμένου τα εργοστάσια να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Και το οποίο μάλιστα αν επιμεριστεί σε κάθε τεμάχιο φτάνουμε σε αυτό το ποσό των 10 cents. Αλλά σας ρωτώ γιατί αυτό δεν έχει γίνει ακόμα εάν τελικά το κόστος ανά τεμάχιο είναι μικρό σε σχέση ιδιαίτερα με το, τη σημασία που έχει αυτό για την βιομηχανία συνολικά. Και τι θα έπρεπε να γίνει για να συμβεί. Πολύ συχνά σε τέτοιου τύπου συζητήσεις έχουμε την αίσθηση ότι το μεγάλο μέρος του κόστους ενός ε, ε, είδους έρχεται από το πολύ χαμηλό κόστος εργασίας. Θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ποιο είναι το ποσοστό του κόστους εργασίας στην τελική τιμή των προϊόντων ρουχισμού. Ναι, βεβαίω ο καταναλωτή μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει λιγάκι παραπάνω, αλλά θα είχε σημασία να γνωρίζουμε και ποιο μέρο ε, της τη τιμή αυτή τελικά είναι το, το ποσοστό κέρδου των εταιριών ρουχισμού. Μιλώντα για βιώσιμη διαρκή αλλαγή, σημαντικό στοιχείο είναι ε, η δυνατότητα των εργαζομένων να οργανώνονται σε συνδικαλιστικούς φορείς και να ασκούν πίεση να ζητούν αξιοπρεπείς αμοιβέ και τήρηση των προτύπων ασφαλείας και υγείας στο χώρο εργασίας. Αναφερθήκατε σε κάποιες αλλαγές στην ενεργοτακή νομοθεσία. Παρόλα αυτά, οι κυβερνητικέ οργανώσει οι οποίε ασχολούνται με το θέμα και εργάζονται επί τόπου έχουν εκφράσει πολλέ ανησυχίε. Για παράδειγμα, περιστολή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντέ, ε, για παράδειγμα τον ελάχιστο αριθμό ε, εργαζομένων που απαιτούνται προκειμένου να συσταθεί σωματείο. Κάτι που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αυτή η δυνατότητα ε, οργάνωσης συνδικαλιστικών φορέων δεν έχει επεκταθεί και στην ε, ειδική ζώνη μεταποίησης προς εξαγωγή που είναι μια περιοχή στην οποία έντονη οικονομική ε, δραστηριότητας. Στο τέλος της προηγούμενου έτους είχαν τεθεί μια σειρά στόχων αριθμητικών για επιθεωρητέ κτλ. Δεν ήθελα να γνωρίσω περισσότερες πληροφορίες για το ποια είναι η πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Για παράδειγμα αυτή η επιπλέον 200 επιθεωρητές στους οποίους αναφερθήκατε επαρκούν δεδομένου του μεγέθους του κλάδου στη χώρα. Και κάτι ακόμα σε σχέση με την ποινική δίαξη, για παράδειγμα του ιδιοκτήτη του κτίριου. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια πρόοδος έχει σημειωθεί. Ευχαριστούμε. Θα περάσουμε στις επόμενες πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Μάρτιν από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πρέσβη. Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας έδωσε και το γεγονό ότι έχουν υπάρξει κάποιες βελτιώσεις. Ε, βέβαια είναι λυπηρό να χρειάζεται να συμβεί μια τόσο μεγάλη τραγωδία για να αντιδράσουμε. Η ανταπόκριση από ορισμένες εταιρείες ηματισμού ευρωπαϊκές ήταν ενθαρρυντική αλλά φαίνεται ότι πιο πολύ τους απασχολεί η εταιρική ε, εικόνα παρά το να αλλάξει η κατάσταση επιτόπου. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την ε, κυρία Πρέσβη να συνεχιστεί η προσπάθεια παρακολούθησης των ενεργειών αυτών των πολυεθνικών εταιριών, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι όντως τηρούν τις υποσχέσεις τους. Ε, δηλαδή, εάν πρόκειται κάτι καλό να βγει από αυτήν την τραγωδία, αυτή η βελτίωση πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη. Δεν μα ενδιαφέρει μόνο τι θα γίνει στου επόμενου λίγου μήνε, αλλά ε, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση και μετά από λίγο καιρό που το ζήτημα θα ξεχαστεί θα επανέλθουμε στα παλιά. Στο θέμα των επιθεωρητών, ζητώ συγγνώμη που θα το πω, μα, αλλά το πρόβλημα στο Μπαγκλαντές, από ό,τι έχω αντιληφθεί, δεν είναι η έλλειψη επιθεωρητών. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από αυτούς τους επιθεωρητές είναι διεφθαρμένοι και χρηματίζονται από τους ιδιοκτήτες των εργοστασίων. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι απλώς να προσληφθούν περισσότεροι επιθεωρητές, αλλά να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και υψηλότερα πρότυπα για τους επιθεωρητές αυτούς. Επίση, θα πρέπει να αυξηθούν οι αμοιβέ αυτών των επιθεωρητών έτσι ώστε να είναι λιγότερο επιρρεπεί στου χρηματισμού. Και υπάρχει και το ζήτημα το ποιο ελέγχει εκείνου που ελέγχουν, να, δημιουργεί ενό ελεγκτικού μηχανισμού. που θα συμπεριλαμβάνει και μια διερεύνηση τη προηγούμενη σχέση που μπορεί να είχαν με του ελεγχόμενους. Αναγνωρίζω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά τα πρότυπα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας, τα πρότυπα στα εργοστάσια ή ακόμα και οι αμοιβέ, δεν θεωρώ ότι μπορεί να επιτευχθεί με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με την ύπαρξη ενός ισχυρού συνδικαλιστικού κινήματος. Επομένω, το επαγγελματία πρέπει να γνωρίζει ότι είναι προ το συμφέρον του ιδίου να υπάρχει συνδικαλισμό, να ε, διασφαλίζονται αυτά τα δικαιώματα στου εργαζόμενου. Και ευελπιστώ να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα. Να διευκρινίσω ότι από την πλευρά μα η σοσιαλιστική ομάδα δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να τιμωρήσουμε το λαό του Μπαγκλαντέ για αυτό που συνέβη, αλλά αντιθέτω να συμβάλλουμε έτσι ώστε η τραγωδία να βοηθήσει. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ. Γιώργος Βαλένσα από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κλωστοφαντουργική βιομηχανία είναι πολύ σημαντική προφανώς ε, και πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας ε, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας ε, για χιλιάδες εργαζομένους. Ακούσαμε ένα κατάλογο δεσμεύσεων σήμερα και χαίρομαι που άκουσα αυτό το κατάλογο και είπατε ότι θα μπορέσετε να εκπληρώσετε τις περισσότερες δεσμεύσεις μέχρι τα τέλη του έτους. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω ποια είναι η πρόοδος, τι έχετε πετύχει μέχρι σήμερα και τι αποτελέσματα μπορείτε να μας παρουσιάσετε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα εδώ. Βέβαια, αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Μπαγκλαντές. Υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα και περιστατικά και σε άλλα μέρη και έχουμε και τις συζητήσεις των ομάδων παρακολουθήσεις για τη βιομηχανία ενδυμάτων και φαίνεται ότι πάρα πολλά πάνε δεν πάνε καλά σε πολλές χώρες και πρέπει να το εξετάσουμε εκ του συνεγγύς. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα τη ευθύνη των εταιριών, κυρίω των ευρωπαϊκών εταιριών, γιατί ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Όταν ευρωπαϊκέ εταιρείε την πηγαίνουν στο εξωτερικό και δημιουργούν ε, τόσο μεγάλα προβλήματα με αποτέλεσμα και θάνατο ανθρώπων. Ε, και ε, χαίρομαι που άκουσα ότι κάποιες εταιρείες ε, θέλουν να συνομιλήσουν, ε, να συμμετέχουν στις συνομιλίες, όμως την περασμένη εβδομάδα στη Γενέβη ε, οι περισσότεροι από αυτούς που είχαν προσκληθεί στις συνομιλίες δεν εμφανίστηκαν καν. Έτσι λοιπόν αυτό εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, τα θύματα εξακολουθούν να περιμένουν για αποζημιώσεις, για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συμβάσεις ε, και αν εταιρείε όπως η Μάνγκο, η Μπένετον και η Βάλμαρτ δεν είναι καν πρόθυμες να συζητήσουν το θέμα και να αναλάβουν την ευθύνη, νομίζω ότι σίγουρα δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα αναγνωρίζουμε τις βελτιώσεις ε, που έχουν ε, γίνει και ελπίζουμε πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες. Ε, θα ήθελα να απευθυνθώ στην πρεσβευτή και να ρωτήσω το εξής. Θα με ενδιέφερε να μάθω τι φόρους πληρώνουν στο Μπαγκλαντές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας πείτε αν καταβάλουν τους φόρους και τι τμήμα του εθνικού προπολογισμού καταλαμβάνουν οι φόροι αυτοί. Επιπρόσθετα, έχει γίνει μια συζήτηση ότι είναι, μεγάλο πρόβλημα, ότι είναι πρόβλημα η υψηλότερη μισθή, γιατί θα υπάρχει μετεγκατάσταση των βιομηχανιών. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτό το επιχείρημα, θεωρείτε ότι είναι σωστό ή ότι είναι ένα ψευδές επιχείρημα που χρησιμοποιείται. Και θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν αν έχετε κάποια διδάγματα και αν σκοπεύετε να αλλάξετε την εμπορική πολιτική προς τα κάποια κατεύθυνση κατόπιν των καταστροφών του Μπαγκλαντές. Επίσης, αν δεν σκοπεύετε να αλλάξετε την κατεύθυνση των εμπορικών πολιτικών, να μας ενημερώσετε και να μας πείτε και γιατί το Κοινοβούλιο έχει δηλώσει ότι θέλουμε να έχουμε δεσμευτικούς κανόνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και νομίζω ότι αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε και πρέπει να δούμε πώς με τις εμπορικές μας συμφωνίες με τις χώρες εταίρους θα διασφαλίσουμε ότι δεν επιβάλλουμε απλώς κυρώσει και αλλά ότι θα βελτιώνουμε και τις συνθήκες εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Και η κυρία Μαρία Μπαντιά από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω εδώ την κυρία Περιβρευτή που περιβρίσκεται εδώ για να μας εξηγήσει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για να αποφευθούν νέες τραγωδίες. Θέλω να τονίσω το όσο υπόθηκαν σε σχέση με την αναγκαιότητα να εμπλακούν ε, όλες οι πληγήσεις οργανώσεις για να βρεθεί μια λύση για την αποφυγή των ατυχημάτων και επίσης να τονίσω την αναγκαιότητα ύπαρξης ανεξάρτητων συνδικάτων. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και να επαγρυπνούν έτσι ώστε οι διαδικασίες σε εφαρμογή χρησιμεύουν. Σε σχέση με τα συνδικάτα θέλω να ρωτήσω αν αυτή η ιδέα εφαρμογής αύξησης των τιμών των προϊόντων αν έχουν τοποθετηθεί σχετικά με το θέμα αυτό το συνδικάτα, αν έχουν γνωμοδοτήσει. Και μια ακόμη ερώτηση σε σχέση με το ψήφισμα του Μαΐου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ένα από τα σημεία ήταν το εξή. Ε, ζητούσαμε την εγγύηση της ε, πλήρους πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη. Έχουν γίνει ε, έχει γίνει κάποια πρόοδο στο σημείο αυτό. Θα σας ευχαριστούσα αν μπορούσατε να με ενημερώσετε σχετικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η συνάδελφος η κυρία Λάμπερτς που είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για την Νοτιοανατολική Ασία βρίσκεται εδώ. Καλώς ορίσατε, θέλετε το λόγο και να συνεισφέρετε στη συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που άργησα. Συμμετείχα σε άλλη συνεδρίαση. Νομίζω ότι μια σειρά από τις παρατήρησεις που έγιναν είναι πράγματι πολύ σωστές. το θέμα των ε, εταιριών που κάνουν τις συμβάσεις, είτε είναι ευρωπαϊκές, αμερικανές κλπ. είναι πολύ σημαντικό, αλλά και αυτό που είπε ο David Martin σχετικά με την ποιότητα των επιθεωρήσεων και του ενδιαφέροντος για το πώ αυτά λειτουργούν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή Απασχόληση έχει ε, μια σχετική ακρόαση αύριο το απόγευμα. Θα ήταν λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τα διάφορα συστήματα επιθεώρηση. Το θέμα χρονοδιαγράμματος ε, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα ήθελα όμως επίσης να μάθω αν υπάρχει πολιτική συμφωνία στο Μπαγκλαντέ μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων ε, όσον αφορά την προώθηση αυτού του θεματολογίου. Γνωρίζουμε ότι σε προεκλογική περίοδο η κυβέρνηση αντέδρασε πάνω στο θέμα αυτό και η ε, ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε πολύ, όπως και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. συμμετείχαν λοιπόν στις συζητήσεις ε, για ένα μελλοντικό σχέδιο. Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει πολιτική συνένεση ώστε άσχετα από το αποτέλεσμα των εκλογών να δούμε να προωθείτε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρινάλντι, ευχαριστώ πολύ. Άλλη από, από, από τους φιλελεύθερους. Ε, Ζητώ συγγνώμη που άργησα, έπρεπε να συμμετάσχω ε, σε συνεδρίαση άλλης επιτροπής. Ε, δεν με εκπλήσει το ότι έχουμε έναν τέτοιο κατάλογο ε, δεσμεύσεων από τις αρχές του Μπαγκλαντές, ούτε με εκπλήσει η καλή πίστη των αρχών του Μπαγκλαντές. Ως μέλος της Επιτροπής όπου προεδρεύει η κυρία Λάμπερτ, πάντα με εντυπωσίασε το υψηλό επίπεδο η πολιτική βούληση ε, της ε, πολιτικής ηγεσία στο Παγκλατές. Και ε, όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε σημαντικές πρόοδους τα τελευταία χρόνια. Τούτου λεχθέντος, συμφωνώ με τον Μάρτιν Ντέιβιτ. Σίγουρα Πέρα από τα νομοθετικά μέτρα υπάρχει και θέμα ανεξαρτησίας ε, του δικαστικού τομέα, ανεξαρτησίας ε, των επιθεωρητών, ανεξαρτησίας ε, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και αυτό αποτελεί πρόβλημα στο Μπαγκλατές. Κάτι που θα απαιτήσει μάλλον μια πολιτιστική διαδικασία, μια διαδικασία που να αφορά την οτροπία, κάτι δηλαδή που ξεπερνάει κατά πολύ τα πλαίσια της νομοθεσίας. Η Φρανσίσκα Κέλλερ ρώτησε σχετικά με τις φορολογικές ε, απάτες. Εγώ θα ήθελα, και εμένα με ενδιαφέρει το θέμα αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ε, πολιτική ε, αποζημίωσης. Η κυρία Πρέσβης εξήγησε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες για να δούμε πώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να αποζημιώσουν τους εργαζομένους ε, υπάρχει γίνονται προσπάθειες για να υπάρχει ε, σωστή νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή, ε, στο ώστε να υπάρχει μια πολιτική αποζημίωση σε, όχι εθελοντική, αλλά να αποτελεί μέρος ενός κώδικα της ε, σχετικής βιομηχανίας, όποτε υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό. Προτού να δώσω το λόγο πάλι στους προσκεκλημένους μας, να τονίσω γιατί βρισκόμαστε εδώ. Δεν ήρθαμε εδώ για να επαναλάβουμε τις συζητήσεις που είχαμε πριν το καλοκαίρι όταν συνέβησαν οι καταστροφές αυτές. Ε, ήρθαμε εδώ για να ελέγξουμε εάν έχει σημειωθεί πρόοδος ε, και αν οι δεσμεύσεις ε, των αρχών του Μπαγκλαντές και των εισαγωγέων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν οι δεσμεύσεις αυτές έχουν ε, ε, επιφέρει αποτελέσματα. Τρία σημαντικά μηνύματα είχαμε στείλει προ του ενδιαφερομένου και τι αρμόδιε αρχέ πριν το καλοκαίρι. Καταρχήν, χαιρόμαστε που το εμπόριο δημιουργεί εκατομμύρια θέσεων εργασία σε φτωχέ χώρε. Είμαστε περήφανοι που η εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι προτιμησιακέ συμφωνίε βοηθούν σε αυτό. Δεύτερον, οι θέσεις αποσχόλησης από μόνες τους δεν αρκούν. Ε, θέλουμε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και στηρίζουμε το πρόγραμμα του Διεθνούς ε, Γραφείου Εργασίας, το οποίο σημαίνει ότι ε, θέλουμε συμμόρφωση με τα πρότυπα παντού. Και Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν θα συνεχίζει να παρέχει προτιμησιακές συμφωνίες σε χώρες που δεν πληρούν ε, τα ελάχιστα πρότυπα. Ο λόγος λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ είναι να ελέγξουμε εάν υπάρχει συμμόρφωση με τις αρχές αυτές. και αν σημειώνεται πρόοδος προς τους στόχους αυτούς. Επόμενος ομιλητής μας ε, είναι ο κ. Φούγκο, ο οποίο εκπροσωπεί το Διεθνέ Γραφείο εργασία. ο οποίος ε, συμμετείχε σε, ε, αποστολή, σε αντιπροσωπεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας υψηλού επίπεδου στο Μπαγκλαντές. Ε, και εξέτασε το σύμφωνο ε, ε, βιωσιμότητας αλλά και άλλα τέτοια θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Λόγκου, από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, Σα ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση. Στόχο είχα να παρουσιάσω μια διακήρυξη, αλλά μέρο των όσων ήθελα να πω τα είπε και η κυρία Πρέσβης. Επιτρέψτε μου, ε, λοιπόν, ε, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω, να δώσω συνέχεια σε αυτά που είπε η κυρία Πρέσβη. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και ποιε θεωρούμε ότι θα είναι οι ε, επικείμενε προκλήσεις. Να ξεκινήσω από τον Ιούνιο-Ιούλιο με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας ε, που υπεγράφει στις 8 Ιουλίου. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο καμπής η πρωτοβουλία αυτή της Κομισιόν δηλαδή. Και θέλουμε να επικροτήσουμε την ε, πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, διότι όλα αυτά ειλικρινά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση του Μαγκλατές, ε, τους κοινωνικούς εταίρους ε, αλλά και την διεθνή κοινότητα να διατηρήσουν ε, την πίεση για να γίνουν ε, οι απαραίτητες αλλαγές. Με το Σύμφωνο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κυβέρνηση πράγματι έχει κάνει πολλά και όπως ε, είπε και γι' αυτό η κυρία Πρέσβης, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αλλαγές στον εργασιακό νόμο. Ο νέος νόμος λοιπόν 15 ε, Ιουλίου αν θυμάμαι καλά ε, εκδόθηκε και ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας εξέδωσε ανακοινοθέν τύπου όπου εκφράζουμε την ανησυχία μας όπως ανέφερε και η κυρία Πρέσβης. Πρέπει να τονίσουμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με το νέο αυτό νόμο. Ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τη Σύμβαση 88 ε, του 98. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο βασικά στοιχεία υπάρχει ε, η απέτηση ε, του ελαχίστου ποσοστού 30% εάν θέλουν οι εργαζόμενοι ε, να δημιουργήσουν συνδικαλιστική οργάνωση. Εάν έχουμε 5.000 εργαζομένους, χρειάζονται 1.500 για να δημιουργηθεί συνδικαλιστική οργάνωση. Πιστεύουμε ότι αυτό το ποσοστό είναι υπερβολικό σε κάποιες περιοχές ε, το ποσοστό ε, στην πραγματικότητα ναι, έρχεται σε 10%. Από την άλλη μεριά όμως, ε, να πω ότι είναι θετικό, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σύμφωνα με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να συνεχίσει να εργάζεται ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αποδεκτά επίπεδα. Η δεύτερη μου παρατήρηση σχετίζεται με ε, την πρόοδο που ανέφερε και η κυρία Πρέσβης. Ε, ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε δύο πράγματα. Καταρχήν, η οικονομική ζώνη, η PZ, να αποτελεί επίσης σε μέρος των συζητήσεών μας και σε συνεργασία με το Γραφείο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στην ΤΑΚΑ να διασφαλίσουμε Ε, να ε, δημιουργηθούν ε, τα διατάγματα, οι κανονισμοί κτλ. που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου. Η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική φάση, το καταλαβαίνετε αυτό. Και Είναι σημαντικοί όλοι αυτοί οι κανονισμοί και τα λοιπά για ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας σε συνεργασία με το IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, περιμένουμε τους κανονισμούς ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Επίσης, θετικό είναι το θέμα της επιθεώρησης. Θα πρέπει να το δούμε αυτό από δύο πλευρές. Έχουμε την επιθεώρηση των κτηρίων που ε, απαιτεί δουλειά μηχανικών και κατόπιν έχουμε την επιθεώρηση εργασίας όπου αναμένεται η πρόσληψη 200 ε, επιθεωρητών. Όσον αφορά την μηχανική πλευρά, ως Ευρωβουλευτές μπορείτε να συνεχίσετε να ασκείτε πίεση σε όλους τους φορείς, ε, ώστε να συνεχίσουν να επιδεικνύουν ε, καλή πίστη στο θέμα του συντονισμού, του καλύτερου συντονισμού. Και επίση έχουμε το θέμα ε, του αισθήματος ιδιοκτησίας, της οικειοποίησης. Η κυρία Πρέσβης είπε ότι ως διεθνής κοινότητα μπορούμε να ε, μπούμε στη χώρα και να διορθώσουμε τα πράγματα σε τρεις μήνες. Αλλά ε, έτσι διασφαλίζουμε μόνο μακρο... βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και ε, το ε, θέμα της οικειοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι ανησυχίες μας συνδέονται με με τα θέματα ε, ε, διαφθοράς, είτε αυτά είναι πραγματικά, είτε ο κόσμος απλά θεωρεί ότι υπάρχουν. Για να χειριστούμε λοιπόν το θέμα αυτό, συνεργαζόμαστε με ένα από τα πανεπιστήμια και δεν προσπαθώ να διαφημίσω το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, αλλά πρόκειται για το ε, Πανεπιστήμιο Μηχανικής και Τεχνολογίας ε, του Μπαγκλαντές. Όταν επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο αυτό τον Μάιο, ε, χάρηκα πολύ που, σε όλη, που υπήρχε γενικά συνένεση σχετικά με την αξιοπιστία του Πανεπιστημίου και, μεταξύ, ε, και, και στη διεθνή κοινότητα και ε, στους ε, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μέρος του προγράμματος μας λοιπόν είναι να συνεργαστούμε μαζί τους για να κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Δεν θα ήθελα να αμφισβητήσω αυτό που είπε η κυβέρνηση, αλλά η επιθεώρηση θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για 3.500 εργοστάσια τα οποία θα πρέπει να επιθεωρηθούν. Και το σύμφωνο που έχει υπογραφεί από τις ευρωπαϊκές μάρκες ουσιαστικά. Υπάρχουν και κάποιες ε, αμερικανικές, ε, αυστραλέζικες και καναδικές εταιρείες επίσης. Αλλά η συμφωνία αυτή θα καλύπτει 1800 με, 1800 2.000 ε, ε, εργοστάσια. Ε, η Αμερικανική Ένωση θα καλύπτει γύρω στα 500 με 500 με 700 εργοστάσια και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας θα πρέπει να καλύψει τα υπόλοιπα. Και στις 7-8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην ΤΑΚΑ σε μια προσπάθεια όλα τα μέρη να χρησιμοποιούν κοινώς αποδεκτά πρότυπα ώστε να αντιμετωπιστούν κάποιες αμφιβολίες ότι τα εθνικά πρότυπα μπορεί να μην αρκούν. Αυτή είναι άλλη συζήτηση, δεν θέλω ε, να μπω στο θέμα αυτό, αλλά το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ η... Ε, δεν είναι τόσο πολύ η ικανότητα ε, επιθεώρησης, είναι το τι αποτελέσματα θα έχουμε από όλα αυτά και τρόπος ώστε να αντιμετωπίσουμε έστω και μερικό στο θέμα είναι τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων να δημοσιεύονται κατευθείαν στο διαδίκτυο. Ε, και επίσης όλοι να είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτά. Ε, τα αποτελέσματα δηλαδή να συζητηθούν στη Διευθύνουσα Επιτροπή που ανέφερε η πρέσβης. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά αναφερθήκατε στις αρχές ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, για την καλύτερη εργασία. Μιλάμε για τον τομέα του ρουχισμού και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε άλλος ομιλητής, ότι το θέμα αυτό ξεπερνάει τα σύνορα του Μπαγκλαντές. Δεν θα πρέπει να έχουμε ε, διπλά μέτρα και σταθμά. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση, την ορμή και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην κατηγορούμε μόνο τον Μπαγκλαντές και να έχουμε ε, δύο μέτρα και σταθμά. Με το νέο εργασιακό νόμο στο Μπαγκλαντές, δυσαρεστηθήκαμε που είδαμε να μην αντιμετωπίσετε επαρκώς το θέμα της παιδικής εργασίας. Επίσης, η αξιολόγηση των κτηρίων πρέπει να ξεκινήσει στο τέλος αυτού του μήνα επαναλαμβάνω αυτό που υπόθηκε. Ε, η Ένωση των Ευρωπαϊκών Εταιριών, λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή προσλαμβάνει προσωπικό, ε, ενώ η Ένωση των Αμερικανικών Εταιριών πραγματοποίησε επίσκεψη αντιπροσωπείας στην ΤΑΚΑ, ώστε να διασφαλίσει την έγκαιρη έναρξη του προγράμματος. Είμαι βέβαιος ότι αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, Ε, θα αρχίσουμε να βλέπουμε αλλαγέ. Επίση, ε, το εμπορικό μα πρόγραμμα, το πρόγραμμα κατάρτιση, συγγνώμη, προβλέπεται να ξεκινήσει αρχέ Οκτωβρίου. Όσον αφορά τα θύματα και τους επιζώντες, Αρκετοί από τους ε, επιζώντες ε, ακροτηριάστηκαν, ε, μπορεί λοιπόν να μην μπορέσουν να ξενεργαστούν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν προγράμματα κατάρτισης ώστε να εργαστούν σε άλλες θέσεις εργασίας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και η Ένωση Εργοδοτών Θα πρέπει να εργαστούν λοιπόν στο νέο πνεύμα, να σεβαστούν ε, το δικαίωμα τους να τι ε, τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα, όσα ανέφερε η κυρία Πρέσβης. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω όλα. Αρκετοί από εσά αναφέρατε ένα πλοκό θέμα, το οποίο είναι το θέμα της αποζημίωσης. Από τον Μάιο και μετά που ήμουν εκεί, Ξέρω ότι η κυβέρνηση ε, έχει αρχίσει να προβλέπει μια αποζημίωση, δεν γνωρίζω το πόσο ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα ξεκίνημα που θα πρέπει να καλύψει τις, ε, κάποιες πρώτες ανάγκες. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αυτή είναι η ελάχιστη αναμενόμενη αποζημίωση. Αυτό είναι κάτι που αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει από μόνη της και το θέμα είναι πώς θα καθορίσουμε το σωστό ποσό. Δεν νομίζω ότι στην νομοθεσία υπάρχει σχετικός κανόνας. Ε, έτσι λοιπόν ζητήθηκε η βοήθεια του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις την προηγούμενη εβδομάδα ε, ανέλαβε πρωτοβουλία να οργανώσει σχετικές συναντήσεις. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα καθορίσει κανείς το ποσό της αποζημίωσης. Έχουμε κάποιες συμβάσει που καλύπτουν τα θέματα αυτά, έχουμε και κάποιους επιρογνώμονες που μας βοηθούν στο θέμα αυτό. αλλά έχουμε και θέμα της κατανομής ε, του βάρου, σε τι ε, ποσοστό θα πρέπει να πληρώσουν ε, οι διεθνείς αγοραστές, οι ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτες του κτηρίου και η κυβέρνηση. κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει σύντομα να οργανώσουν ε, συνάντηση οι πολυεθνικές εταιρείες ε, για να εξετάσουν το θέμα. Επίσης, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι μας πιέζει ο χρόνος, να κάνω μια έκκληση, ε, κάτι που ανέφερε και ένας από τους προαλαλήσαντες. Όπως είπε η κυρία Πρέσβης, το θέμα αυτό είναι θέμα ανάπτυξης. Ναι, το, Διεθνές, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ενδιαφέρεται για την απασχόληση και τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά είναι θέμα ανάπτυξης. Θα χρειαστεί βοήθεια λοιπόν η χώρα για να καθορίσει το επιχειρηματικό μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη, όπως πολύ σωστά είπατε, το συγκριτικό πλεονέκτημα ε, για το που έχει το Μπαγκλαντές, ε, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική παρέμβασή σας. Θα ήθελα όμως να σας απευθύνω μια ερώτηση. Λαμβάνοντας υπόψη το ζήτημα της πολιτικής βούλησης της υιοθέτηση νομοθεσίας, της εφαρμογής της νομοθεσίας, της αποτελεσματικής ε, εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Από αυτές λοιπόν τις απόψεις πώς θα εκτιμούσατε την κατάσταση, ποια είναι τα ε, σημεία στα οποία οι αρχές του Μπαγκλαντέ θα έπρεπε να εστιάσουν περισσότερο, προς ποια κατεύθυνση θα έπρεπε και εμείς ίσως να πιέσουμε. Ποια είναι λοιπόν τα αδύναμα σημεία σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ ότι το θετικό στοιχείο είναι ότι γρήγορα υιοθετήθηκε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ε, ήταν κάτι που συζητήθηκε, ένας νόμος που συζητήθηκε τέσσερις φορές, ήταν κάτι που ε, επέδειξε πολιτική βούληση ο Πρωθυπουργό ε, και πίεσε τα μέλη της κυβέρνησης. Λοιπόν, υπήρξε πρόοδος εκεί. Στην εξάλληψη των ε, περιορισμών στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε, Οι ειδικοί του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας το έχουν εξετάσει από τεχνικής απόψεως και είναι σημαντική η πρόοδος. Μια άλλη σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στο επιχειρησιακό πεδίο. Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια επιτροπή η οποία πραγματικά εργάζεται. Συνεργάζεται με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και άλλους φορείς και με ένα τρίο ας πούμε πρέσβης της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών και της, ε, της Ολλανδίας. Και κάθε ε, εβδομάδα γίνεται μια συνάντηση αυτή τη Επιτροπή, συνεργασία με την κυβέρνηση για να δουν πώς πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια. Αυτά ήταν θετικά. Τώρα πηγαίνοντας σε μια στα, στα πιο αδύναμα σημεία είναι τα εξή. Το ερώτημα του κατά πόσον αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο και αυτά τα νέα μέτρα θα μπορέσουν να υιοθετηθούν πριν τις εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο, απολύτως απαραίτητο για να προχωρήσουμε. Εσείς το γνωρίζετε ως βουλευτές καλύτερα από μένα ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας νόμος αν δεν υπάρχει σχετική βούληση. Αμέσως μετά τις εκλογές λοιπόν θα πρέπει να επανέλθουμε στο ζήτημα αφενός του 30% για τη σύσταση συνδικαλιστικού φορέα και αφετέρου στο ζήτημα της ε, ζώνης μεταποίησης προς εξαγωγή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ε, αυτό το ποσοστό το 30% το θεωρώ υπερβολικά μεγάλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ε, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και την άποψη των Ευρωπαίων ενδιαφερόμενων φορέων. γιατί νομίζω ότι και οι φορείς αυτοί ε, υπέστησαν συνέπειες από αυτήν την τραγωδία. Ξεκινώ από τον κύριο Φραντσίσκο Μάκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ξεωτιμοί ε, βουλευτές, ξεοτιμή κυρία Πρέσβη. Σας ευχαριστώ που καλέσατε τον φορέα μας που εκπροσωπεί τον ευρωπαϊκό τομέα της κλωστοϊφαντουργίας με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόθεση της κλωστοϊφαντουργίας στην Ευρώπη. Εκπροσωπούμε 180.000 εργασίες, ε, εταιρείες ε, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό στην Ευρώπη και πολλές από αυτές είναι μικροπισές επιχειρήσεις. Εδώ και 15 χρόνια η Eurotext έχει υπογραμμίσει τη σημασία της υιοθέτηση και και του σεβασμού προτύπων σε ολόκληρη την κλωστοϊφαντουργία και στην αλυσίδα εφοδιασμού της βιομηχανίας αυτής. Αυτό είναι απαραίτητο για την εικόνα και την αξιοπιστία της βιομηχανίας μας και επίσης για τη διασφάλιση ενός ισότιμου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους για να δημιουργήσουμε, για να οργανώσουμε προγράμματα ευαισθητοποίηση στον τομέα τη εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδιαίτερα σε συνεργασία με μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά και παγκοσμίω. Σε σχέση με το Μπαγκλαντέ, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι το 2010 εισήγε η Ευρώπη 8,5 δισεκατομμύρια τεμάχια αιματισμού από τη χώρα αυτή. Είναι η δεύτερη χώρα σε εισαγωγές μετά την Κίνα. Η χώρα αυτή έχει ωφεληθεί, όπως σωστά αναφέρατε, από το πρωτομισιακό καθεστώς. Είναι μία από τις λίγες χώρες που αυξάνει το μερίδιο αγοράς της. Πέρυσι και μάλιστα και φέτος αυτή η αύξηση του μεριδίου αγοράς συνέχισε παρά την ε, κρίση. Αλλά ε, είναι σαφές ότι οι περισσότερες από αυτές τις αγορές προέρχονται από ευρωπαϊκές εταιρείες είτε και παρόλο που μερικές φορές χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι. Και υπάρχει ένα ζήτημα διαφάνειας εδώ. Πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε ότι το τραγωδία στο Ράνα Πλάζα δεν σταμάτησε το εμπόριο. Οι εμπορικές συναλλαγέ με τον Παγκλαντές αυξήθηκαν σε όγκο 6,6% και δεν υπάρχει κανένα αίσθημα ε, αλλαγής της ε, τάσης αυτής. Από τη στιγμή υπάρχουν συμβάσεις, αυτές θα τηρηθούν. Το ερώτημα είναι πώς. Ας είμαστε ξεκάθαροι, από τη δικιά μας την πλευρά, είμαστε ιδιαίτερα, ε, θεωρούμε ιδιαίτερα τραγικό τα γεγονότα στον Μπογκλαντές, αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτό καθιστά τη χώρα ξεχωριστή. Δυστυχώς, αυξάνονται τα τέτοιου τύπου εργατικά ατυχήματα σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ασία. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι τα διεθνώ αποδεκτά πρότυπα δεν εφαρμόζονται. Την πλευρά του φορέα μας λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι. Το Μπακλαντές δεν είναι η μόνη χώρα η οποία αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Επιτρόπου Ντεγκούχτ και όλες τις άλλες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε επίπεδο Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες μέσω διμερών επαφών για τη βελτίωση της κατάστασης. Η συμμετοχή της κυβέρνησης και των αρχών της χώρας είναι κρίσιμη σημασία, καθώς επίσης και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα όμως από την πολιτική υποστήριξη και την οικονομική βοήθεια, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να ε, αποδώσει προτιμοσιακό καθεστώς σε μια χώρα, θα πρέπει να διασφαλίζονται ε, σεβαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή δίνονται αυτά τα προτιμησιακά καθεστώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν ευθύνη να εξετάζουν και να διασφαλίζουν ότι οι χώρες αυτές υιοθέτησαν και τηρούν και πληρούν τα κριτήρια. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή κατά την άποψή μας. Να μην ακολουθούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Συμφωνώ και εγώ με πολλούς από τους προλαλήσαντες ότι δεν πρέπει να ε, χαθεί αυτή η κινητικότητα που έχει ξεκινήσει τον Ιούλιο στη Γενέβη ο Φερές μας εκπροσωπήθηκε για να υποστηρίξει το σύμφωνο. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή είναι καλύτερη από την ε, πρόταση των Βόρειο Αμερικανικών ε, της Αμερικανικής ε, Συμμαχίας Κλωστοϊφαντουργίας, αλλά ο τομέας της κλωστοϊφαντουργίας παραμένει ιδιαίτερα κατακαιρματισμένος. Ο έλεγχος βρίσκεται ακόμα στα χέρια των ε, εταιριών λιανικού εμπορίου και ακόμα περισσότερο ε, των ε, εταιριών διανομής. Ειλικρινά σας λέω ότι δυστυχώς μόνο εξαιτία αυτού του τραγικού ατυχήματος και της δημοσιότητας που έλαβε, ξεκίνησαν αυτές οι πρωτοβουλίες και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα σταματήσουν. Πολλές από τις εταιρείες δεν θα έλεγα ότι περίμεναν το ετύχημα για να κάνουν κάτι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν αυτές οι εταιρείες να ελέγξουν τα πάντα. Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να ε, ελέγξουν την κατάσταση στους προμαθευτές τους στο εξωτερικό. Προφανώς υπάρχει κόστος στην τήρηση αυτών των προτύπων, αλλά αυτό το κόστος δεν μπορούμε να το βάλουμε στην ίδια ζυγαριά με το, τις ανθρώπινες ζωές και εγώ αγοράζω ρούχα, αλλά δυστυχώς τελικά οικονομικά κριτήρια επικρατούν, γι' αυτό ο δρόμος θα συνεχίσει να είναι μακρύς. Καλωσορίζω την προσπάθεια να μην ε, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις πρωτοβουλίες και να υπάρξει καλύτερο συντονισμός. Μόνο έτσι οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μπορούν να γνωρίζουν με σαφήνεια ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Όπως σωστά ελέγχθη όλες οι σχετικές συμφωνίες 4-3-4 εστιάζουν σε ορισμένα από τα σημαντικά θέματα. Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε ε, και παραπέρα Λοιπόν, αυτή τη διαδικασία η οποία θα είναι διαρκής και θα γίνει φηματικά θα μπορέσουμε να περάσουμε σε άλλα ζητήματα πέρα από τα προφανή στο τομέα αυτό. Οι εταιρείε που εκπροσωπεί ο φορέας μας δεν σταμάτησαν τις δραστηριότητές τους μετά το ατύχημα. Ορισμένες δραστηριοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, όπως ε, για παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου υπάρχει συνεργασία με την κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πολλές από αυτές τις εταιρείε ανέλαβαν πρωτοβουλίες χωρίς μεγάλη δημοσιότητα, ανταποκρινόμενες στις ε, συμφωνίες που ε, συνήφθησαν στη, στη Γενέβη. Και, ε, υπογραμμίζω το ατύχημα στον Παγκλαντές είναι τραγικό, αλλά δεν είναι μοναδικό. Τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν και σε άλλα μέρη του κόσμου. Πρέπει λοιπόν το ζήτημα της του πρωτομεσιακού καθεστώτος να το εξετάσουμε συνολικά και επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να επισημάνω ότι σε αυτήν εδώ την Επιτροπή θα συζητηθεί το ζήτημα του GSP Plus και ποιες χώρες θα ε, συμμετάσχουν. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για την Επιτροπή και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει την αποτελεσματική τήρηση κοινωνικών, ε, ε, περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων τήρησης σεβασμού των δικαιωμάτων. Η διαδικασία αυτή διαρκεί, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, όχι μόνο για τον Παγκλαντές, αλλά για οπουδήποτε στον κόσμο. Η Eurotex θα συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους για την ε, προώθηση προγραμμάτων που αυξάνουν τον σεβασμό του περιβάλλοντος και τον σεβασμό των ε, κοινωνικών ε, δικαιωμάτων και θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην ξεχνούν ότι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να επιτρέψει αλλά και να ενθαρρύνει τις ε, ευρωπαϊκές πλωστοϊφαντουργίες να παράγουν προϊόντα τοπικά. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σα για το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων ΣΥΝ. επενθυμίσω στο κριτήριο ότι οι απαιτήσει ε, για τη συμμόρφωση με το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων ΣΥΝ είναι πολύ πιο απαιτητικέ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει το αν αυτές οι απαιτήσει πληρούνται από όσου ζητούν συμμετοχή στο σύστημα αυτό να σας θέσω μια ερώτηση. Τα μέλη της ε, Ένωσής σας που έχουν υπογράψει το σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν να συστήσουν κάποιο μηχανισμό για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να έχετε μια εποπτεία σχετικά με το αν συμμορφούνται τα μέλη σας. Θα είμαι ε, μαζί σας, Πρόεδρε. Αν δείτε τον ε, οριθμό των μεγάλων εταιριών ε, που έχουν ε, υπογράψει το σύμφωνο με το Μαγκλεντές είναι περιορισμένος ο αριθμός των πολυεθνικών και οι περισσότερες, αν όχι το 99%, είναι κυρίως εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε λιανικό επίπεδο. Μεταξύ των μελών μας, θέλουμε τώρα να διασφαλίσουμε ότι μικρές και μεσές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό θέτουν πρόσθετα ερωτήματα. Παραδείγματο χάρη σε σχέση με τα πρότυπα ασφαλεία ή τι συνθήκε εργασία, τα πρότυπα εργασίας. Όμως αυτά όλα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο εταιρεία. Ε, ήθελα να είμαι ειλικρινή μαζί σα, γι' αυτό σα απαντώ έτσι. Μέχρι σήμερα για μας αυτό είναι ένα θέμα εταιρικό. Επιμένουμε να εφαρμόζουν τα μέλη μας σωστά τα ελάχιστα πρότυπα και δεν υπάρχει αντίρρηση για αυτά τα ελάχιστα πρότυπα. Το αντίθετο, πολλά μέλη μας πηγαίνουν και παραπέρα. Και ξέρω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, υπάρχουν κάποιες ενώσεις που συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις σε επίπεδο κράτους μέλους για να βελτιώσουν την κατάσταση όταν παραδείγματο χάρη συνεργάζονται με τον Μπουγκλέτε, αλλά και όχι μόνο. Και το τονίζω αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και επίτηδε, ο ε, τελευταίο ομιλητή θα είναι ο Κόρτσιμπετ ο οποίο ε, εκπροσωπεί την Ένωση Ελευθερού Εμπορίου και κυρίω ε, τους εισαγωγείς ενδυμάτων σε επίπεδο λιανικής δεν είναι μυστικό ότι έχει τεθεί η ένωσή σας ε, στο στόχαστρο. Τι έχετε να πείτε για τις κατηγορίες αυτές που έχουν ακουστεί εναντίον σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, κύριε Αναπληρωτή και Διευθυντή, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ ε, το λιανικό εμπόριο έχουμε περίπου 1150 εταιρείες ε, μέλη μας και οι περισσότερες έχουν ε, συμμετάσχει στο μηχανισμό βελτίωσης, παρακολούθησης και βελτίωσης της κοινωνικής συμμόρφωσης των εταιριών. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι καταρχήν ότι αυτές οι εταιρείες εισαγωγής ε, ουσιαστικά εκπροσωπούν πολλές πολυεθνικές, αλλά εμείς εκπροσωπούμε πέρα από τις πολυεθνικές και πολλές μικρές και μεσέ επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη γκαμετεριών που εισάγουν προϊόντα όχι μόνο από τον Μπαγκλαντές, αλλά και από όλο τον κόσμο και επίσης, όπως είπαν και οι γίνεται γίνονται πολλέ συζητήσει τώρα για τον Μπαγκλαντέ και βεβαίω συμφωνούμε ότι πολλά πρέπει να γίνουν στον Μπαγκλαντέ και ανησυχούμε όλοι τα μάλα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις μεγάλες τραγωδίες που είδαμε στο τεστριν στην Ράνα ε, Πλάσα αλλά και σε άλλα εργοστάσια και κάτι πρέπει να αλλάξει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπογραμμίσω ότι πρέπει να σκεφτούμε και τι συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες όπου βλέπουμε παρόμοιες προκλήσεις. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις ε, ολιστικά. Καθολικά δεν θέλουμε να δακτυλοδείξουμε μια συγκεκριμένη χώρα, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς δικούνται οι επιχειρήσεις στην παγκοσμία λυσίδα. Έτσι λοιπόν η FTA έχει δημιουργήσει την BSAI και νομίζω όλο και περισσότεροι γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό κρόνιμο. Έχουμε τρει πυλώνε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει και στον Μπαγκλαντέ αλλά και σε άλλε χώρε. Κίνα, Ινδία, σε πολλέ άλλε χώρε. Το πρώτο στοιχείο αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης ε, στην ε, αλυσίδα προμήθειας ε, και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και πολλές έχουν τονιστεί. Έχουμε το θέμα της ελευθερίας, ε, του συνεταιρίζεστε, των μισθών, ε, των συνδικών εργασίας, αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά για να κάνουμε μια αλλαγή, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, το ζωτικό είναι να έχουμε μια βελτίωση. Γι' αυτό τακτικά οργανώνουμε πάρα πολλά workshop κατάρτιση σε όλο τον κόσμο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και για να εξηγήσουμε πώς οι διευθυντές των εργοστασίων μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο που εργάζονται. Γιατί δυστυχώς εξακολουθούν πολλοί να πιστεύουν πως όταν μιλάμε για την ε, κοινωνική συμμόρφωση αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον αγοραστή ή τον ελεγκτή όχι εδώ μιλάμε για σεβασμό των κανονισμών, για σεβασμό της νομοθεσίας των παγκλεντές, για να μιλάμε για το σεβασμό των συμβάσεων ε, της ΔΟΕ, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ε, και ελπίζουμε ότι όλες ε, οι εταιρείες κατά μήκος της Ελσίδας σέβονται τα μέτρα αυτά. Παρ' όλα αυτά, επίσης βλέπουμε ότι ο, τρόπο, ο δρόμος προς την εφαρμογή αυτών των προτύπων είναι πολύ μακρύς. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα. Και αν πράγματι θέλουμε να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες για να το πετύχουμε αυτό και να δούμε βελτιώσεις και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, βήμα το βήμα μικρές ε, βελτιώσεις, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Όλα αυτά θα τα πετύχουμε μόνο αν εργαστούμε όλοι μαζί. Και οι αγοραστές και τα εργοστάσια και οι εμποριλιανικείς και οι ε, ενώσεις των επιχειρήσεων, οι κυβερνητικές αρχές, τα συνδικάτα, η Ακαδημαϊκή Ένωση Βιομηχάνων, Εξαγωγείων Ενδυμάτων του Μπαγκλαντέ. Δεν έχει νόημα να δεκτυλοδεικνούμε ένα στον άλλο και να λέμε «Άσε, δεν έχει κάνει τη δουλειά σου καλά, εμεί την κάναμε καλύτερα». Όλοι μαζί πρέπει να εργαστούμε επί του αυτού, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να σημειώσουμε την αλλαγή. Και προκειμένου επίση να διευκολύνουμε ένα διάλογο για τα θέματα αυτά στι κύριε χώρε πηγή, και ιδιαίτερα στον Μπαγκλαντές έχουμε ξεκινήσει κάποιες στρογγυλές τράπεζες που λαμβάνουν χώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να βρούμε και ενδυνάμει λύσεις. Όμως το σημαντικό είναι διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη στα διάφορα επίπεδα να συνομιλήσουν και όχι να διαφωνούν, γιατί το είδαμε αυτό σε κάποιες χώρες. Έτσι λοιπόν σε τοπικό επίπεδο όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η τοπική δικαιοποίηση και εμείς το πιστεύουμε αυτό σε αυτή. Γιατί αν δεν υπάρξει ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο τότε δεν θα πετύχουμε. Δεν θέλω τώρα να επαναλάβω επί των διάφορων πρωτοβουλειών ε, που έχουν αναλυφθεί από διάφορες εταιρείε ε, και από συνδικάτα, η Accord Alliance, ορισμένα μέλη της FTA και η BSEI έχουν συνυπογράψει τις συμφωνίες σε σχέση με τη βελτίωση της ασφάλειας στο Μπαγκλαντές. Ε, καλωσορίζουμε αυτή την κίνηση πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για να κινηθούν τα πράγματα και βασίζεται στο διεθνές τριμερές σχέδιο δράσης που νομίζουμε ότι μπορεί να επιφέρει τις αλλαγές τις οποίες επιζητούμε επεγνωσμένα. Όμως, η μόνη ανησυχία που βλέπω σε σχέση με αυτές τις διάφορες πρωτοβουλίες είναι ότι υπάρχει ένας κίνδυνος επικαλύψεων. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε πώς αυτές οι διάφορες οδοί ανάληψης δράσης είναι συντονισμένες και να αποφύγουμε την επικάλυψη, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει και σύγχυση και κούραση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που πρέπει να έχουμε κατά νου. Είναι σημαντικό να προσθέσω το εξή. Πιστεύουμε ότι το Μπαγκλαντέ επίση βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ευχαρίστω θα υποστηρίξουμε και τα ενδιαφερόμενα μέρη του Μπαγκλαντέ ε, για να καταλήξουν σε μια επιτυχή έκβαση. Εμείς ε, δεν θέλουμε να κινηθούμε σε άλλες αγορές, ως αγοραστές, ε, ως Θέλουμε να προμηθευόμαστε από τον Μπαγκλαντές και στο μέλλον. Αυτό είναι σαφές. Έχουμε εργαστεί με προμηθευτές από τον Μπαγκλαντές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν εξελίξεις προς την ορθή κατεύθυνση και θέλουμε να συνεχίσουμε. Και αν άλλοι επιλέξουν άλλες αγορές, τότε αυτό δεν θα ωφελήσει τον κλάδο ούτε τη χώρα. Λεχθέντων αυτών, Νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολλά θέματα, χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο, αλλά θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην πρόοδο σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο στον Παγκλατές και αναλαμβάνουμε και τη δική μας ευθύνη, έχουμε μερίδιο της ευθύνης και αναμένουμε και περαιτέρω καρποφόρες συζητήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον Παγκλατές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω μία παρατήρηση και να θέσω μία ερώτηση. Η παρατήρηση, κατα, καταρχάς. Πώς αντιδράτε στην κατηγορία που ακούστηκε επανειλημμένα εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις τραγωδίες του Μπαγκλαντές. Ότι δηλαδή τα μέλη σας εποφελήθηκαν περισσότερο από ε, τις ε, κακές συνθήκες εργασίας ε, και τους χαμηλούς μισθούς στο Βαγγλαντές. Μετά από το σύμφωνο που υπέγραψαν τα μέλη σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχετε κάνει για να συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεώσεις. Έχετε δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης της συμμόρφωσης με αυτές τις υποχρεώσεις. Ναι. Υπάρχει υποχρέωση για τις εταιρείε που συμμετέχουν στο PSCI. Αυτό δεν αφορά μόνο το Μπαγκλατές, είναι ε, κάτι, είναι υποχρεώσεις ε, τις οποίες ε, υποχρεούνται να τηρούν τα μέλη μας σε όλες τις χώρες. Και παρακολουθούμε τα εργοστάσια, τις κοινωνικές συνθήκες και εάν οι επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες, ε, τις διώχνουμε από την ε, Ένωση αυτήν, κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας βέβαια, αλλά το κάνουμε επειδή θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Γίνονται και διαφανείς αναφορές στο θέμα αυτό στην ετήσια έκθεση. Δεν είναι λοιπόν κρυφά όλα αυτά και πρέπει να ομολογήσω ότι πολλά από τα μέλη μας σε πολλά από τα μέλη μα δεν αρέσει αυτό ή κατά κάποιο τρόπο είμαστε εμεί η αστυνομία, αλλά αν δεν κάναμε κάτι τέτοιο δεν θα ήμασταν πια αξιόπιστοι. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσεί πώ βλέπετε την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να πάρω το λόγο σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και ε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω μετά από τόσους διακεκριμένους ομιλητές. Ε, ε, προέρχομαι από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Κομισιόν και το Μπαγκλαντές είναι πολύ καλό παράδειγμα για μας και της σημασίας του εμπορίου για την ανάπτυξη και της σημασίας σημαντικών εγχώριων πολιτικών για να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη για το λαό. Αναφερθήκατε στη σημασία του, ε, της βιομηχανίας ρουχισμού για τον Μπαγκλαντές και των ευρωπαϊκών εισαγωγών. Μιλάμε για 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ ε, πέρσι, ε, κάτι που αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕΠ της χώρας και νομίζω ότι μπορούμε να υπολογίσουμε ότι 2,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ε, σχετίζονται με αυτό. Το Μπαγκλαντές επωφελείται από ε, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς ε, δασμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον τομέα έτοιμου ρουχισμού. Το γεγονός ότι το Μπαγκλατές καλύπτεται από την Γενική Συμφωνία, από το Γενικό Πρωτομησιακό Πλαίσιο, ε, μας δίνει και μια ευκαιρία να ενεργήσουμε, διότι έτσι έχουμε μια ειδική σχέση ε, και δυνατότητα για διάλογο ε, καθώς και επιπλέον κανάλια επικοινωνίας σε δύσκολες περιστάσεις. Πουθενά νομίζω δεν ακούστηκε τόση αλληλεγγύη όσο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από του καταναλωτέ, από ε, συνδικαλιστικέ οργανώσει, από εργοδότε και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Επιτροπή ΙΝΤΑ, διότι ε, είχατε σημαντικό αντίκτυπο στα όσα ε, ακολούθησαν. Το Μπαγκλαντέ δεσμεύτηκε να βελτιώσει τι συνθήκε εργασία και ασφαλεία ε, στα εργοστάσια μετά από το σύμφωνο που υπογράψαμε με την κυβέρνηση του Μπαγκλατές και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ε, Οι Ηνωμένε Πολιτείε κατόπιν συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια ε, συνεργαζόμαστε και με ενδιαφερομένους. Ε, η συμφωνία αυτή είναι κυρίως ε, διακυβερνητική, ε, δεν συνυπογράφουν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ. Να σας πω πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό. Το σύμφωνο αναφέρει δύο ειδών αποτελέσματα, τα βραχυπρόθεσμα, ε, την ε, δυνατότητα του συνεταιρίζεστε και άλλα εργασιακά πρότυπα, η υιοθέτηση ε, κατάλληλων κανόνων εφαρμογής. Αυτό αναφέρθηκε ως πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς και να αναφέρω επίσης την πρόσληψη 200 επιθεωρητών εργασίας. Κατόπιν έχουμε πιο ε, μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα να πω μεσοπρόθεσμες ε, δεσμεύσεις ε, που συμπεριλαμβάνουν ε, να επεκταθεί ο εργασιακός νόμος και για τις οικονομικές ζώνες μεταποίησης και επικροτούμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση για τις προσπάθειές της και για την τροποποίηση του νόμου. Αφήνουμε στο Διεθνές Γραφείο Εργασία να αξιολογήσει την τροποποίηση αυτή του νόμου. Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά ε, σημάδια. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ε, δεδομένων των περιορισμών ε, που υπάρχουν στην αναπτυσσόμενη αυτή χώρα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αναλάβει μια σειρά δράσεων μέχρι το τέλος του χρόνου και παρακολουθούμε στενά την ε, ε, την πραγματοποίηση αυτών των δεσμεύσεων. Πολύ πιο σημαντικό είναι ότι και ο λαός του Παγκλαντές ε, παρακολουθεί την κατάσταση. Σύντομα θα πραγματοποιηθούν εκλογές, όπως και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές παρακολουθούν την κατάσταση. Και αναφέρθηκε το πώς μπορούν οι καταναλωτές να, παίξουμε, να παίξουν ρόλο αγοράζοντας υπεύθυνα. Τέλος, έχουμε τη Διευθύνουσα Επιτροπή του Διεθνού Γραφείου Εργασίας και την Εργασιακή Διάσκεψη που θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά ε, την κατάσταση στο Μπαγκλατέ, ε, διότι τα συμπεράσματα ε, των σχετικών φορέων μας ενδιαφέρουν και στα πλαίσια εμπορικών συμφωνιών όπως είναι η συμφωνία τα πάντα εκτός από όπλα, everything but arms. Επίσης στο σύμφωνο ε, αναφέρθηκε η ημερομηνία του 2014 ως ορόσημο για την ε, παρακολούθηση της πρόοδου, αλλά οι επόμενοι μήνες θα είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να γίνουν πραγματικές αλλαγές ε, στη χώρα και θα ήθελα να αναθαρρύνω την κυβέρνηση του Παγκλατές να συνεργαστεί στενά με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για να επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Επιτρέψτε μου και να απαντήσω σε μια ερώτηση που τέθηκε από κάποιον Ευρωβουλευτή, νομίζω, από τους πράσινους ε, σχετικά με το αν η Επιτροπή σκοπεύει να αλλάξει την εμπορική πολιτική της ε, ε, μετά από τα γεγονότα στο Μπαγκλαντές. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσω ότι φυσικά συνεχώς επικαιροποιούμε την εμπορική πολιτική μας και θα γνωρίζετε ότι πριν ένα χρόνο εκδώσαμε ανακοινωθέν σχετικά με τα με θέματα εμπορίου και είδαμε ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε την εμπορική μας πολιτική ε, ε, ώστε να ακολουθεί τις εξελίξεις. Η εμπορική πολιτική είναι μόνο μία πλευρά ε, του όλου θέματος. πιο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστούν και άλλες πτυχές ώστε η ε, εμπορική πολιτική να είναι βιώσιμη. Ε, το αίσθημα ιδιοκτησίας, ε, οικιοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι εγχώριες πολιτικές, αλλά και ο ρόλος μας ως διεθνής εταίροι είναι πολύ σημαντικός. Και υπάρχει το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ε, το πώς μπορούν ε, να ενσωματωθούν τα θέματα αυτά στην εμπορική πολιτική μας. Έχουμε λοιπόν ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου νέας γενιάς όπου υπάρχουν σαφείς αναφορές στα διεθνή μέσα που αφορούν την εμπορική κοινωνική ευθύνη όπως είναι ε, ο σχετικός αμερικανός, ε, αμερικανικός κώδικας για το θέμα αυτό. Και επίσης, όσον αφορά το GSP και το GSP+, ε, το πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών. Αυτά είναι μέσα που παρέχουν κίνητρα και μας επιτρέπουν να έχουμε συζητήσεις με τις διάφορες χώρες σχετικά με τη βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων ε, κλπ. Μια δυνατότητα που δεν θα είχαμε αν δεν συμμετείχαν στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω και δημοσίως ότι προσωπικά ε, εκτιμώ τη στάση που τήρησε η Επιτροπή ως εκτελεστική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ε, ε, σαφής ξεκάθαρη η στάση της και απέτησε από τα αποτελέσματα. Και προφανώς ο Επίτροπος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Μπορούμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας δίνοντας το λόγο στην πρέσβη του Μπαγκλαντές. Ξεχότατη. Κυρία Πρέσβη, έχετε το λόγο. Μήπως θα προτι... Όχι, ο πρόεδρος διευκρινίζει ότι στο τέλος θα μιλήσουν οι βουλευτές. Κύριε Πρόεδρε, λέει η πρέσβη, δεν εννοούσα ότι θα έχω εγώ τελευταία κουβέντα. Προφανώ τα μέλη του Κοινοβουλίου θα έχουν την τελευταία ε, κουβέντα. Λοιπόν, προσωπικά πρέπει να πω ότι βρήκα ιδιαίτερα διαφωτιστικές και ενθαρρυντικές ορισμένες από τις ερωτήσεις που μου ετέθησαν ε, και κάποιες από τις παρατηρήσεις από τον αναπληρωτή ε, Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ...την εκπρόσωπο της Eurotext, καθώς επίσης τον εκπρόσωπο των εταιριών κλιανικού εμπορίου και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορισμένα από τα ερωτήματα που έθεσαν οι βουλευτές μετά την παρουσίασή μου θεωρώ ότι ε, ως έναν βαθμό έχουν απαντηθεί από τις ε, τοποθετήσεις που ακολούθησαν σε σχέση για παράδειγμα με τους επιθεωρητές όπως ε, ξεκαθάρισα δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ομάδα εργασία που θα ασκεί αυτούς τους ελέγχους αλλά και μια Αμερικανική και άλλες. βρισκόμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού. Ε, χτες μόλις βρέθηκαν στην ΤΑΚΑ οι ε, επιθεωρητές από την ε, Βορειοαμερικανική Συμμαχία. Και υπάρχει μια προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των Αμερικανικών και των Ευρωπαϊκών ε, ελεγκτών για να μην υπάρξει αλληλοεπικάλυψη. Να μην βρεθούμε σε καταστάσεις στις οποίες για παράδειγμα ξαφνικά αυτές οι, και οι τρεις αρχές θα πήγαιναν να ελέγξουν ένα εργοστάσιο αυτό θα σημαίνει ότι θα έπρεπε να σταματήσει η παραγωγή εκεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάρτιν για τις παρατηρήσεις του. Αναφερθήκατε ε, στο ζήτημα της ε, ποιότητας του ελεγκτικού μηχανισμού και όχι τόσο του αριθμού των ελεγκτών. Όπως είπε και ο πληρωτής Γενικός Διευθυντής του ILO, συμμετέχει το Πολυτεχνείο του Μπαγκλαντές σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης που έχει ιδιαίτερα καλή φήμη ε, και θα ασκήσει αυτούς τους ελέγχους. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εμπιστοσύνης το ζήτημα της διαφθοράς είναι παγκόσμιο και ας είμαστε καλόπιστοι, ας θεωρήσουμε ότι δεν είναι όλοι οι ελεγκτές διεφθαρμένοι. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η ορμή, αυτή η κινητικότητα, όχι μόνο από την πλευρά του Μπαγκλαντές, αλλά και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, εταιριών λιανικού ε, εμπορίου, της Eurotex. Όπως ανέφερε και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα γίνουν την επόμενο έτος συναντήσεις για αξιολόγηση της προόδου και απολογισμού. Ε, αναφέρθηκε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο στο Μπαγκλαντές και αυτό δημιουργεί ζητήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων και των προτύπων ε, στο χώρο εργασίας θα εγκαταλειφθεί ή θα ξεχαστεί. Όλα τα πολιτικά κόμματα μαζί ε, ε, έχουν συμφωνήσει, τους ανησυχεί το θέμα, έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους στο Κοινοβούλιο Και αυτό νομίζω ανταποκρίνεται και στην απέτηση του λαού να υπάρξει πραγματική αλλαγή και όχι απλώς λόγια. Γιατί, όπως σωστά είπε και η εκπρόσωπος της Επιτροπής, το θέμα είναι ότι ο λαός του Μπακλαντές μας παρακολουθεί. Εάν είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις εφημερίδες, τον τύπο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Μπακλαντές θα διαπιστώνατε το τεράστιο ενδιαφέρον και το πόσο πολύ βρίσκεται στο στόχαστρο ο τομέας της κλωστοϊφαντουργίας για προκειμένου να ε, υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία, πρέπει να δημιουργηθούν συμβιβασμοί, ε, να υπάρξουν συμφωνίες μεταξύ των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και ας μην ξεχνούμε επίσης και τους εισαγωγείς, την πλευρά εκείνη της εφοδιαστικής αλυσίδας που καταλήγει στις εταιρείε γενικού εμπορίου. Ε, κύριε Μέρφυ, ρωτήσατε ποιο είναι το ποσοστό του εργατικού κόστους. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, δεν γνωρίζω το ακριβές ποσοστό. αλλά θέτω το εξής ερώτημα. Πληρώνουμε μια τιμή για ένα ρούχο σε ένα κατάστημα εδώ. Ποιο ποσοστό αυτής της τιμής είναι το κόστος. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και εδώ είναι το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μπορεί να αυξηθεί η πίεση, μπορεί να αυξηθεί η πίεση από την κοινωνία των πολιτών ε, ή από την διεθνή κοινή γνώμη. Ο τύπος έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία παρακολουθώντας και ε, φωτίζοντας την τραγική κατάσταση στον Μπακλαντές μετά, τις, μετά δύο ατυχήματα. αλλά θα ήθελα να δω την ίδια δημοσιότητα και προσοχή από την πλευρά του τύπου και προς τους άλλους. Έτσι ώστε και εκείνοι να συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις. Αυτό το συμπέρασμα αντλώ από την συνάντηση στη Γενέβη την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν από την πλευρά του το Διεθνές Γραφείο εργασία και μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να προσελκύσουν τις εταιρείε παραγωγή ρούχων, εννιά ήρθαν. Αυτό κάτι μας λέει νομίζω. Και αυτές οι εταιρείε είναι απρόθυμες να αναλάβουν το κόστος της αποζημίωσης ρίζονται. Το επιχείρημά τους είναι γιατί εμείς πρέπει να αναλάβουμε το κόστος ενός ατυχήματος στην ΔΑΚΑ. Αυτό είναι ε, απογοητευτικό γιατί πρόκειται για ένα είδος υπεργολαβίας, outsourcing. Αυτές οι εταιρείε με την έδρα τους για παράδειγμα στην Ευρώπη δίνουν υπεργολαβίες σε εταιρείε στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς, για παράδειγμα στην πληροφορική, για παράδειγμα τα τηλεφωνικά κέντρα, όταν ε, μια αεροπορική εταιρεία, για παράδειγμα, διατηρεί το τηλεφωνικό της κέντρο στο, σε χώρα της Ασίας. Δεν θα με κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πιστεύω ότι τα διεθνή μέσα μαζική ενημέρωση θα έπρεπε να εστιάσουν και σε αυτό. Δεν λέω ότι εμεί από την πλευρά μα το Παγκλαντέ δεν έχει ευθύνη, αλλά πρέπει να δούμε το ζήτημα τη ετορική και κοινωνική ευθύνη και από αυτήν την πλευρά. Εάν θέλουμε να μην επαναληφθούν τέτοια ατυχήματα που έχουν τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό κόστο για το Πακλαντέ, μα πηγαίνει πολλά βήματα πίσω στην ανάπτυξη και είναι και μια ανθρωπιστική καταστροφή τελικά. Και θα ήθελα να έχω διαβεβαιώσει από τους εταίρους μας σε αυτή τη διαδικασία, από εσά από την ILO, από τι μη οργανώσει από του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, από τους προσώπους των εταίριων. Και αν είχα αυτές τις διαβεβαιώσεις θα τις διαβιβάσω στην ΤΑΚΑ. για να γίνουν αυτές οι διαβεβαιώσεις πράξη. ετέθησαν και άλλα ζητήματα. Θα ήθελα για παράδειγμα να απαντήσω στην κυρία Κέλλερ ε, που ανέφερε το ζήτημα της φορολογίας των ευρωπαϊκών ε, εταιριών. Ε, δεν έχω τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Μέρφυ ξέχασα να πω ότι ε, εκπρόσωπος Κομισιόν ήταν η Μόνικα Χέτζετ από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΤΡΕΙΤΟ. Ο κύριος Μέρφυ, ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Ε, κάποια σχόλια που τα εμπνεύστηκα από τις εμπνεύσεις ε, της Eurotex και της FTA. το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ κακές ε, συνθήκες εργασίας στην κλωστοφαντουργία στον Παγκλαντές δεν είναι κάτι καινούριο σίγουρα. Είχαμε κάποιες τραγωδίες τους τελευταίους μήνες, ε, τα είδαμε στην πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όμως δεν πρόκειται και κάτι καινούριο, δεν αποτελεί έκπληξη. Τα ήξεραν ε, οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα και το γεγονός ότι συμβαίνει και σε άλλες χώρες δεν αποτελεί δικαιολογία για να μην αναλάβουμε δράσεις σε σχέση με τα εργοστάσια που σχετίζονται με το Μπαγκλαντές. Ε, όμως, ε, όπως σας είπα, δεν είναι μεμονωμένη η κατάσταση στο Μπαγκλαντές και δεν είναι κάτι καινούριο και πρέπει να δούμε ότι το Μπαγκλαντές παράγει για όσο δυνατό μικρότερο κόστος όσο είναι δυνατόν και αυτό σημαίνει ότι δεν σέβεται τους κανονισμούς για τις πυρκαγιές, τις συνθήκες εργασίας και τις ε, τα πρότυπα ασφαλεία. Και αυτό δεν έγινε κατά λάθο κάποιοι ωφελούνται από αυτό και εγώ νομίζω ότι πρέπει να απορρίψουμε ότι αυτοί που κερδίζουν είναι οι καταναλωτέ στη Δύση αλλά αυτοί που κερδίζουν είναι όσοι κερδίζουν από τη φύση αυτή του κλάδου και έχουμε δει πάρα πολλές εκθέσεις αν διαβάσετε κάποιε συνεντέύξει γίνεται αναφορά στο ε, πόση μεγάλη δύναμη έχουν μεγάλοι αγοραστές εισαγωγείς ε, και τα καταστήματα λιανικής. Αυτοί φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη εξουσία και επομένω έχουν ευθύνη για το τι συνέβη, αλλά έχουν και ευθύνη σε σχέση με την αλλαγή. Και νομίζω ότι το πραγματικό ερώτημα, ερώτησε ο πρόσωπος του FTA, το εξή, αν οι εταιρείε που εκπροσωπούνται από την FTA θα επέλεγαν να πάνε σε μια άλλη χώρα, αν το Μπαγκλαντές ε, δεν εφαρμόζει όσα έχουν ε, συμφωνηθεί σε σχέση με τις επιθερήσεις εργασίας ε, κτλ. Και αν συμβαίνει κάτι θα χρειαζόταν μια περίοδος χρόνου. Όμως εγώ νομίζω ότι η πιο σημαντική ερώτηση είναι αν η τιμή των ενδυμάτων, αν ανέβαινε 10 λεπτά του ευρώ ανά τεμάχιο, και ακούσαμε ότι αυτό είναι το κόστος για να βελτιώσουμε τα πρότυπα ασφαλείας, τότε στο στάδιο αυτό θα μετακινούνταν σε άλλη χώρα όπου δεν θα υπήρχε αυτή η αύξηση των 10 cents και ίσως να το έκαναν και τότε στη συνέχεια δεν θα διονυζόταν αυτό το πρόβλημα σε άλλη χώρα. Έχουμε λοιπόν ε, το, το θέμα ε, του τι συμβαίνει στον Μπαγκλαντές ε, θα μπορούσε πραγματικά χάρη να μετακινηθούν οι εταιρείε να μετακομίσουν αλλά νομίζω ότι τα θέματα παραμένουν τα ίδια. Έχουμε το θέμα λοιπόν ε, της αμοβολής, μια διαδικασία επεξεργασίας που γίνεται στον Μπαγκλαντές εγώ νομίζω πάντως ότι αν ε, υπήρχε αυτή η αύξηση δεν θα άρεσε στην FTA γιατί μάλλον αυτό θα σήμαινε περικοπή του κέρδους. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας. Ε, νομίζω ότι ήταν πραγματικά παραδειγματική η συζήτηση που έχει να κάνει με το πώς πρέπει να βλέπουμε την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη διασυνοριακή ροή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά δεσμευόμαστε από το Σύνταγμα για να ενδιαφερόμαστε για τα κοινωνικά πρότυπα. Ελπίζω λοιπόν να στεφθεί με επιτυχία η περίπτωση του Μπαγκλαντές και τελικά να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι εμείς είμαστε τμήμα της λύσης και φέρνουμε καλύτερες θέσεις και ασφαλέστερες θέσεις εργασίας στον Μπαγκλαντές και αλλού. Λοιπόν, να περάσουμε στο σημείο 28. Πρόκειται για την τροποποίηση του κανονισμού 2173 του 2005 του Συμβουλίου για τη δημιουργία εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για εισαγωγές ξυλίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όπως ξέρετε, το FLEGT σημαίνει για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και διαχείρισης για την ξύλια. Υπάρχουν ε, άλλες αξίες λοιπόν εδώ που πρέπει να διαφυλάξουμε. Εμεί είμαστε η αρμόδια επιτροπή. Η είναι ο κύριος Βίγκλερ από το ΕΛΚΑ. Θα αντικατασταθεί από το Χέρος Κλαβαλένσα από την ίδια πολιτική ομάδα και θα του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορεί να παρευρεθεί ο κ. Βικλέρ σήμερα. Έτσι λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, θέλω να διαβάσω την δήλωση που έχει προετοιμάσει ο Οργανισμό του Συμβουλίου 73 του 2005, καθιερώνει σύστημα αδειών για την επιβολή τη δασική νομοθεσία, διακυβέρνηση και εμπόριο, φέρει τα αρχικά φλεκτ. Αυτό το σύστημα στοχεύει στην αντιμετώπιση τη παράνομα λειτουργούμενη ξυλία και του συναφού εμπορίου εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα ξυλίας που προέρχονται από κάποιες χώρες εταίρους, δηλαδή χώρες που έχουν συνάψει εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει των παραμέτρων αυτών ορίζει ότι μόνο προϊόντα ξυλίας που έχουν ε, υλοτομηθεί νόμιμα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία σε αυτές τις χώρες εταίρους μπορούν να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν ε, δεν υπάρχει άδεια εισαγωγή FLECT, η εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ξυλίας από τις χώρες εταίρους απαγορεύεται. Η πρόταση που εθετήθηκε από την Επιτροπή δεν στοχεύει στην τροποποίηση των ουσιαστικών χαρακτηριστικών του συστήματος ενδιών ΦΛΕΚΤ στοχεύει στην ε, προσαρμογή των διατάξεων επιτροπολογίας του κανονισμού για το σκατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή και άλλες προτάσεις ε, ευθυγράμμισης ανέμεναν ε, το θετικό αποτελέσμα των διοργανικών διαπραγματεύσεων Omnibus 1 και 2, καθώς καταλήγουμε στη συμφωνία για τα Omnibus, μπορεί να προχωρήσει η εργασία σε άλλους φακέλους. Ε, ο προτινόμενο τροποποίηση του κανονισμού ε, χωρί την Επιτροπή την εξουσία να υιοθετεί και εκτελεστικέ ε, πράξεις και κατεξουσιοδότηση πράξη. Πρόταση δίνει στην Επιτροπή την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικέ πράξεις σύμφωνα με τον κανονισμό 182 του 2011 για να αξιολογήσει και να εγκρίνει τα εφιστάμενα συστήματα που ε, διασφαλίζουν ε, την ε, ανείχνευση των προϊόντων ξυλίας που εκφράζουν από τις χώρες εταίρους. Αυτό μπορεί να αποτελέσει λοιπόν την βάση για τις άδειες φλέκτα. Αυτά τα συστήματα σήμερα αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Τροπολογίας υπό την κανονιστική διαδικασία. Η πρόταση δίνει στην Κομισιόν την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις συγγνώμη, ε, της πράξης σε σχέση με την εξαίρεση των προϊόντων ξυλίας των ειδών που προηγούνται στα τρία παραρτήματα του κανονισμού 338 του 97 για την προστασία ειδών άγρια πανδέ και χλωρίδα. Δεύτερον, την υιοθέτηση κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού FLECT που ρυθμίζει την πρακτική λειτουργία των συστημάτων άδεια εισαγωγών και τρίτον τροπολογίες στο παράρτημα 1, 2 και 3 του κανονισμού FLECT που, όπου αναφέρονται οι χώρες και τα προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα διοδότησης σε σχέση με τις εκτελεστικές εξουσίες. Ο κύριος, Βίνκλερ, έχει προτείνει μια τροπολογία που θέλει να διασφαλίσει ότι τέτοιες εξουσίες ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 182 του 2011 στο σύνολό του, παρά σύμφωνα μόνο με το άρθρο 5 του κανονισμού σε σχέση με τις κατεξουσίες της πράξης, ο κ. Βίγκλερ έχει προτείνει δύο τροπολογίες. Καταρχήν, ε, για τον κύριο Βίκλερ, η διάρκεια της εξουσιοδότησης ε, δεν πρέπει να είναι αόριστη. Αντιθέτως, θα πρέπει να περιορίζεται στα πέντε έτη με σιωπηρή, αυτό με τη σιωπηρή επέκταση. Παράταση. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων Omnibus 2, επομένως πρέπει να το σεβαστούμε. Δεύτερον, ο κύριος Βίγκλερ θεωρεί πως οι τρεις τομείς όπου η εξουσιοδότηση θα δοθεί ε, πρέπει να υποτελεί στοιχείο πολιτικής ευχέρειας. Έτσι λοιπόν η περίοδος αντίρρησης για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι δύο μήνες με τη δυνατότητα περαιτέρω παράτασης τεσσάρων μηνών και όχι δύο. Αυτό αντικατοπτρίζει την, ε, το σκεπτικό των συμφωνιών ε, Omnibus 1 και 2 για το θέμα αυτό. Και πάλι θα πρέπει να αποφύγουμε αποκλήσεις. Αυτά προετοίμασε για μένα, Επομένω περιμένω και τι δικέ σα απόψει. Μάλιστα, άρχεται η συζήτηση, λέει ο πρόεδρο. Ε, καταρχήν ο κ. Ζεντό από πράσινου. Πράσινους. Ευχαριστώ. Γενικά, συμφωνούμε επί της έκθεσης με τον εισηγητή και κυρίως σε ό,τι αφορά τις της πράξης. Όμως έχω μία διπλή ερώτηση για το άρθρο 1 την απευθύνω στον εισηγητή και ίσως και στην Κομισιόν. Έχουμε μία εξέλιξη για το θέμα της αναγνώρισης ε, των ετικετών, των label, για να αιτιολογούμε την άδεια FLECT. Και υπάρχει μία εξέλιξη που φαίνεται σοβαρά ουσιαστικά να αποδυναμώνει τις ετικέτες που θα μπορούσαν να γνωριστούν. Έχουμε τις διεθνείς ετικέτες FSE και είναι σοβαρές και έχουν καλή φήμη και ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές ετικέτες είναι ενδιαφέρουσες σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό δάσος, όμως ε, αντιθέτως ε, ε, υπάρχουν κάποιες ετικέτες που τοπικά αμφισβητούνται. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το διακύβημα, υπάρχει μια εξέλιξη στο κείμενο και θέλουμε να ξέρουμε γιατί. Και το δεύτερο σημείο αφορά το θέμα της ανιχνευσιμότητας. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό στα πλαίσια του ΦΛΕΚΤ για να μπορούμε να ελέγχουμε την νομιμότητα της ξυλίας, της εισαγόμενης ξυλίας. Και εδώ προτείνεται ε, να περάσουμε σε εκτελεστικές πράξει για την ανιχνευσιμότητα. Εμεί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να μείνει σε κατεξουσιοδότηση πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Μία επιπλέον ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Κατεξουδότηση πράξης για τροποποίηση του κανονισμού με προσθήκη επιπλέον χωρών κτλ. Η Κομισιόν προβλέπει να προσθεθούν ε, ξεχωριστά οι χώρε με διαφορετικές κατεξουδότηση πράξεις ή με μία κατεξουσιοδότηση πράξη ε, μπορούν να καλυφθούν διαφορετικές χώρε. Διότι αυτό φυσικά επηρεάζει την ε, ικανότητα του Κοινοβουλίου να ελέγχει τα πράγματα αυτά. Ευχαριστώ. Ακούσαμε ερωτήσεις. Λογικέ ερωτήσει, αλλά δεν είναι εισηγητή. Αλλά είμαι βέβαιο ότι θα μεταφερθούν στον εισηγητή οι ερωτήσει αυτέ Να ρωτήσουμε την Κομισιόν. Μπορεί να μα απαντηθούν οι ερωτήσει. Ποιο είναι παρόν. Τρία ονόματα έχω. Yes. Name for the record, please. Το όνομά σας παρακαλώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Σβετλάνα Ετενάσοβα από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Η πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού FLECT είναι πολύ απλή, όπως ήδη αναφέρθηκε. Δεν έχει στόχο ε, καμία ουσιαστική τροποποίηση του κειμένου θα πρέπει να θεωρηθεί μια απλή ευθυγράμμιση του κανονισμού με την ε, πραγματικότητα ε, που ισχύει τώρα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν περιμέναμε λοιπόν ερωτήσεις που να αφορούν την ουσία του κανονισμού αυτού. Σας ευχαριστούμε όμως για αυτές. Ευχαριστώ. Θα απαντήσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση. Ε, την τροποποίηση των κανονισμών. Όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε δει ακόμα να υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση των ε, παραρτημάτων, ε, διότι δεν είχαμε καμία εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέσης. Το σύστημα θεωρείται ότι λειτουργεί καλά. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που χρειάζεται τροποποίηση κάποιο παράρτημα του κανονισμού. Πόσο σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσες συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή πόσα συστήματα εντός αυτών των ε, συμφωνιών ε, θα ε, καταστούν λειτουργικά. Δεν θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε την τροποποίηση κάποιου παρατήματος ε, εάν ε, ισχύει κάποια θελοντική συμφωνία εταιρική σχέσης ε, και είναι έτοιμο το σύστημα να τεθεί σε λειτουργία. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να τροποποιήσουμε τα παρατήματα εάν βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Εάν θεωρηθούν ε, λειτουργικά ε, πάνω από ένα τέτοια συστήματα, μπορούμε να σκεφτούμε να τα χειριστούμε ως πακέτο. Ένας από τους στόχους μας ε, όμως, και αυτό μάλιστα είναι και ένα από τα επιχειρήματά μας, που ζητάμε να είναι δύο συν δύο μήνες το διάστημα ε, που μπορεί να υποβάλει αντίρρηση στο Κοινοβούλιο αντί για το αρχικό 2 συν 4 μήνες. Ε, ε, ένα από του λόγου λοιπόν είναι να μπορούμε να αντιδράσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε περίπτωση τροποποίησης κάποιας διεθνούς συμφωνίας ή συμφωνίας εταιρική σχέσης. Μόλις λοιπόν έχουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι ικανό να εκδίδει πιστοποιητικά φλεκτ, θα πρέπει να μπορέσουμε και εμείς ε, να τροποποιήσουμε γρήγορα την εσωτερική μας ε, νομοθεσία στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, το σήμα ΦΛΕΚΤ, που ουσιαστικά το ονομάζουμε επιστοποιητικό ΦΛΕΚΤ, Είναι ένα θέμα το οποίο δεν πιστεύαμε ότι θα ξανασυζητήσουμε. Έχει συζητηθεί επανειλημμένα η αξιοπιστία του συστήματος. Καθορίζεται με τον κανονισμό του ΦΛΕΚ. Γενικά το σύστημα θεωρείται αρκετά στεναρό ώστε να μπορεί να ε, παρουσιάζει αποτελέσματα. Θεωρείται αξιόπιστο. Πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη και ποια θα είναι τα αποτελέσματα τη στιγμή που θα εκδοθούν πιστοποιητικά φλέκτα. Αυτό ε, θα το δούμε, διότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία αποδείχθηκε πιο ε, πολύπλοκη από ό,τι περιμέναμε από την αρχή. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Τανάσοβα. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν στόχο έχει ευθυγράμμιση του κανονισμού με το νέο καθεστώς ε, και εκτελεστικών πράξεων. Ε, ο εισηγητής δέχεται ε, ε, τους περιορισμούς της εντολής της Κομισιόν. Ας δούμε αν άλλα μέλη της Επιτροπής μας θα ξεπεράσουν τα όρια αυτά. Ο εισηγητής προτείνει δύο τροπολογίες. Να υπάρξει περιορισμός ε, της εξουσιοδότησης. κάτι συνηθισμένο από την πλευρά του Κοινοβουλίου και προβλέπει και παράταση του, ε, της προθεσμίας ε, για υποβολή αντιρρήσεων. Ε, τίποτα νέο λοιπόν. Ας δούμε τι θα αποφασίσουμε κατά την ψηφοφορία. Ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 24 ε, του μήνα, 6 το απόγευμα. Προβλέπεται ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας, στην κανονική μας συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τέλος του δημοσίου μέρους της συζήτησής μας σήμερα. Το, η συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και κλεισμένων των, των θυρών. Παρακαλώ λοιπόν ε, όσους δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν για το και κλεισμένων των θυρών κομμάτι της συνεδρίασης να εγκαταλείψουν την ε, αίθουσα όσο γίνεται πιο